Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά. Στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ για την, παρουσία σας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να χαιρετήσω την Δήμαρχο της Λαμπεντούσα, την συνάδελφο κυρία Νικολίνη, την οποία καλωσορίζω θερμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Νικολίνη, νομίζω ότι χωρίς υπερβολή μπορεί να πει κανείς ότι είσαστε όχι μόνο η αρμόδια πολιτικός στο νησί, αλλά και σαν άνθρωπος, αλλά και ως εκπρόσωπος των συμπολιτών σας στην Λαμπεντούζα είσαστε ένας φάρος σε δύσκολες εποχές. Με πολύ σεβασμό και θαυμασμό παρακολουθούμε τους ανθρώπους στο νησί σας ε, και βλέπουμε την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν εδώ και χρόνια. Γνωριζόμαστε πολύ καλά εγώ είχα την ευκαιρία δύο φορές να επισκεφτώ την Λαμπετούζα και είδα πως έχει η κατάσταση επιτόπου. Θα ήθελα λοιπόν όχι μόνο να σας καλωσορίσω, αλλά να σας ευχαριστήσω ε, από καρδίας για τη δουλειά που κάνετε εκεί. Είναι μεγάλη μου τιμή να καλωσορίσω και τον ε, υπεύθυνο της επιχείρησης ε, uniform Med, ε, τον ε, Ναύαρχο Κρεντεντίνο καθώς και τον ε, Ναύαρχο τον υπονάβαρχο Μελώνε που βρίσκεται μαζί μας εδώ σήμερα, καθώς και τους συναδέλφους σας που θα μας δώσουν σήμερα πληροφορίες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εικόνα σχετικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζεται και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ε, η Ιταλία. Επίσης, ε, ο Τζουζέπε Λάι, πληρχός της ε, Φρεγάτας, που ήταν και στο λιμάνι της Λασπέτσια. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και σας θερμά. Αγαπητοί Ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πέρα από ε, τα εισαγωγικά μου λόγια θα ήθελα να πω στην κυρία Νικολίνη ότι επανειλημμένα είχα τη δυνατότητα να βρεθώ σε σκάφος ε, Ιταλικό να δω τη δουλειά που κάνει το πλήρωμα. Επισκέφτηκα επίσης το αρχηγείο σας και ζητώ συγγνώμη που δεν γνωρίζω ακριβώς ε, την ονομασία, αλλά ε, στην Δυτική Σικελία. Μπόρεσα έτσι να συνομιλήσω με τους συναδέρφους σας. Και το έχω πει αυτό και στον Τζόρτζο ε, Ναπολιτάνο και στον κύριο Ματαρέλο. Το είπα και στη Ρώμη, στον, ε, στο ε, αρχηγείο αμήνης. Συνήθως το, το ναυτικό ε, έχει να κάνει με την άμυνα. Ποτέ όμως, και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, δεν είδα τέτοια ανθρωπιστική ε, προσπάθεια όσο αυτήν ε, που ε, είδα από την πλευρά του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Είδα την αφοσίωσή τους, την την βοήθεια που προσέφεραν στους ανθρώπους δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς αυτό και όταν κάποιος είναι ναυτικός σίγουρα, όταν είναι ε, σίγουρα έχει κάποια εικόνα. Αν δείτε όμως τι κάνουν πραγματικά αυτοί οι στρατιώτε ε, οι ναυτικοί για την ειρήνη, μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν είναι μόνο συγκινητικό. Ε, είσαστε τιμή για τη χώρα σας και με αυτά που κάνετε υπερασπίζεστε τα ιδανικά της Ευρώπης. Είμαστε περήφανοι για αυτά που έχει κάνει το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό στη Μεσόγειο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε μπροστά σας τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Ε, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν ε, εάν δεν υπάρξουν ε, αντιρρήσεις στο μεταξύ. Και επίσης... Πρωτού προχωρήσουμε στην ανταλλαγή απόψεων και ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους μας, ε, ζητώ συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας ε, που πρέπει ε, να να πούμε κάποια διαδικαστικά. Στις 22 Οκτωβρίου θα είναι η επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στην Ρώμη. 22 Οκτωβρίου στη Ρώμη. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών θα συναντηθεί στην ε, Βαρκελόνη και ε, η τρίτη ε, συνεδρίαση υψηλού επίπεδου για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για την... Όσον αφορά την ε, συνεδρίαση του Προεδρείου της 11ης Ιουλίου, όπου ε, με εκπροσώπησε ο ε, συνάδελφος Σασόλη, θα ήθελα να σας προτείνω στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης ε, να εξετάσουμε τα συμπεράσματα της συνεδρίασης τη 11 η Ιουλίου. Κατόπιν έχουμε την ομάδα εργασίας ε, για ε, το θεματολόγιο και με την... Υπό την προεδρία της συναδέλφου Πεκίν, η ομάδα εργασία συνεδρίασε στις 29 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προχωρήσουμε πάλι στο βασικό θέμα Τη σημερινή ε, ημερήσια διάταξης που είναι οι ανθρωπιστικές προκλήσεις ε, που συνδέονται με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Θα ήθελα κυρίε και κύριοι να δώσω κατευθείαν το λόγο να προχωρήσουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια. Äh, και πάλι Είδαμε αύξηση των ε, σκαφών ε, όπου πρέπει να σώσουμε τους επιβάτες ε, και έχουμε ένα πρόβλημα κατανομής το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις προσπάθειες που καταβάλλετε εσείς να σώσετε ανθρώπους, οι προσπάθειες που γίνονται για να καταχωριστούν οι άνθρωποι αυτοί, οι προσπάθειες για να εξεταστούν ε, οι περιπτώσεις ε, του καθενός. Äh, äh, äh, και έτσι χαίρομαι που έχουμε ανθρώπους μαζί μας ε, σήμερα που μπορούν να μας πούν πώς έχουν τα πράγματα και προτείνω να ξεκινήσουμε από την κυρία Νικολίνη και κατόπιν ε, να δώσω το λόγο στους ε, δύο αντιναβάρχους. Έχουμε προβλέψει ε, ο καθένας να κάνει μια σύντομη εισαγωγική παρέμβαση και κατόπιν να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Παρακαλώ, κυρία Νικολίνη. Ε, Γεια σας. Ευχαριστώ που ήρθατε και με τιμά η παρουσία σας. Σύντομα να σας παρουσιάσω την κατάσταση που ισχύει στην Λαμπεντούζα και που γνωρίζετε. Έχουμε μια ροή που δεν σταματάει και που οδηγεί σε κύματα μεταναστευτικά που ακολουθούν τα κύματα της θάλασσας τα ίδια. Έχουμε κάποια έτσι και ξαφνικά μας ήρθαν 10.000 άτομα με πολλά παιδιά και γυναίκες αλλά και 30 θύματα. Είχαμε την 1η Οκτώβρη, την 3η επέτειο του Μεγάλου Ναυαγίου, το 2013, και δυστυχώς το γιορτάσαμε αυτό με κι άλλους νεκρούς στη θάλασσα. Αυτή λοιπόν η η ροή είναι ασταμάτητη, όπως ασταμάτητη είναι και η νεκρή και τα ναυάγια. Θα δείτε ο υπονάβαρχος μας έφερε ένα βίντεο που γυρίσαμε στη Λαμπεντούζα για τη σημασία της διάσωσης. Έχουμε να κάνουμε ένα σιωπηλό πόλεμο που δεν σταματάει ποτέ. 11.400 είναι νεκροί από την επέτειο αυτή το 2013 όταν γονάτισε ο ίδιος ο Μπαρόζο εκεί στη Λαπεντούζα και είπε να σταματήσουν οι νεκροί στη Μεσόγειο φτάνει πια και μόνο το 16 είχαμε 3.500 νεκρούς είναι πραγματικά καταθλιπτικό το να παρακολουθεί κανείς όλο αυτό στην Λαμπεντούζα που είναι η μόνη ανοιχτή πόρτα. Η μόνη ανοιχτή πόρτα στον κόσμο και στον Νότο και από φέτος είναι ανοιχτή και προς τον, τον Βορρά γιατί ήρθαν και γύρω στους 400 νέους να γιορτάσουν μαζί μας αυτή την επέτειο μαζί με τους μετανάστες που επιβίωσαν. Εκεί θα δείτε τον κόσμο να κλαίει όταν καταθέτει τα λουλούδια στον τόπο του ναυαγίου. Και βλέπουμε όμως ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το πιο σημαντικό που θέλω να σας πω εγώ εδώ είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Αλλιώς ο αριθμός των νεκρών δεν θα σταματήσει ποτέ. Ένα άλλο τρόπο να μιλήσει κανεί για τη Λαμπεντούζα είναι το να μιλήσει και για τι θετικέ πλευρέ. τη διασώση ή και την προβολή τη διεθνή ε, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, μουσικούς, ένας από τη Συρία που έκανε ένα event μουσικό στη, στο νησί. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονται θαμένοι κάτω στη θάλασσα είναι και νέοι με πολλές προσωπικές ιστορίες, όνειρα. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα δεινά του πολέμου. Και αυτό το φοβερό που συμβαίνει τώρα βλέπω πάντως να είναι πιο ευιστοποιημένη η γνώμη και να έχει σταματήσει αυτό και να έχει πέσει λίγα για αυτό το τείχος της Ομπερτά. Ίσως χάρη και στη Λαπεντούζα αυτό ίσως αρχίζουμε να βάζουμε στην άκρη τον εθισμό. Υπάρχει μεγάλη συγκίνηση, κλαίμε μπροστά τις εικόνες των νεκρών μωρών, μπροστά στα ναυάγια, αλλά δεν, κατα, δεν καταφέρνουμε ή δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βοηθήσουμε όπως πρέπει τους ζωντανούς. Πρέπει να τονίζουμε πάντοτε ότι αυτή οι αριθμοί που ακούμε συνέχεια δεν ξέρω κατά πόσο είναι αριθμοί που μπορεί να διαχειριστεί η πυρός μας. Αυτό πάντως που ήρθα να σας πω σήμερα και που είναι σημαντικό είναι ότι μετά το 11 όπου η Λαμπεντούζα ήταν θέατρο προπαγάνδας εισβολής μετά από την Αραβική Άνοιξη στην Τινησία κυρίως. Η Λαμπεντούζα λοιπόν σιγά σιγά άρχισε να και τον τουρισμό τη το 2013 το 2014. Φέτος είχαμε έκρηξη τουρισμού. Αυτό μου φαίνεται το πιο σημαντικό να σας μεταφέρω. Γιατί αποδείξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την έκτακτη ανάγκη, ότι μπορούμε να διοργανώσουμε διάσωση για την υποδοχή χωρίς να πλήξουμε τις τοπικές κοινότητες. Και όχι μόνο. Αποδείξαμε ότι ο τουρισμός αυξάνεται. Η Λαμπεντούζα είναι ένα νησί που ξεπέρασε μια εικοσαετία μεγάλης μοναξιάς. Γιατί ό,τι έκανε Λαμπεντούζα μέχρι την άναξη της επιχείρησης Μαρενόστρουμ τα έκανε μόνη της. Και όχι μόνο δεν χαθήκαμε, αλλά μεγαλώνουμε. Είμαστε ένα νησί με μέλλον και συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε ζωντανούς και δυστυχώς και νεκρούς. Από το Εθνικό Ναυάγιο έχουμε 30 θύματα. 30 σωροί που θα φτάσουν. Σε ένα τόσο μικρό νησί. Αλλά πώς τα πετύχαμε όλα αυτά. Τα καταφέραμε νικώντας την σιωπή και, την, και μέσω της κινητοποίησης όλων των αρχών. ΟΤΑ, δομές υγείας, πολιτών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όχι μόνο της τοπικής κοινότητας αλλά και των τουριστών και της ίδιας Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μεγάλη προπαγάνδα σε σχέση με το σποτάκι αυτό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αν κάποιος αρνείται είναι συμβαίνει επειδή έχουμε το Δουβλίνο όχι επειδή είναι εγκληματίες δεν ξέρω τι άλλο και οι Ευρωπαίοι δυστυχώ δεν έχουν θέσει εφαρμογή το σχέδιο μετακατάστασης και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δυστυχώς αποθούν προς την Ιταλία το διπλώσιο αριθμό των ατόμων που καταφέραμε εμείς οι ίδιοι να μεταγκαταστήσουμε Και αυτό είναι απαράδεκτο. Αν δεν αρχίσουμε λοιπόν να αποδεικνύουμε στους ίδιους τους αυτούς μας σε αυτές τις μικρές περιοχές, τις μεθοριακές που επέδειξαν δύναμη και θάρρος ότι μπόρεσαν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους με σημαντικά στοιχεία. Εμείς ε, στα δύο χρόνια καταφέραμε να μετεγκαταστήσουμε 36.028 ώρες, ενώ δεχτήκαμε 400.000. Πώς γίνεται εγώ και οι άλλοι κάτοικοι της Λαπεντούζα και οι πολίτες της Ευρώπης, πώς γίνεται να έχουμε όλοι εμείς εμπιστοσύνη και να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρώπης. Ελπίζω η δουλειά που κάνουμε στη Λαμπεντούζα να αποβεί χρήσιμη όχι μόνο για μας, όχι μόνο για αυτούς που υποδεχόμαστε, όχι μόνο για τους τοπικούς, για την τοπική κοινότητα, αλλά ελπίζω η Λαμπεντούζα να μην μείνει η μόνη ανοιχτή πόρτα για την Ευρώπη. Γιατί αυτή η ανοιχτή πόρτα είναι μια ανοιχτή πόρτα για το μέλλον. Δεν είναι ανοιχτή πόρτα προς μια εισβολή. Είναι μια ανοιχτή πόρτα προς τη ζωή και το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Νικολίνη. Προτείνω να δώσουμε τώρα το λόγο στους εκπροσώπους ε, του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρώτα στον ε, υπονάμβαρχο Μελώνε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας ζητήσω να μετακινηθούμε για να δούμε πρώτα το φιλμάκι.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 Μήπως γίνεται να έρθει κάποιος τεχνικός να μας βοηθήσει γιατί δεν έχει συνδεθεί ο προτζέκτορας με τον υπολογιστή.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 δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ προτζέκτορα και υπολογιστή.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 Θεωρώ σημαντικό να δείτε αυτό το φιλμάκι επειδή πιστεύω ότι οι εικόνες αξίζουν πάνω από χίλιες λέξεις. Αυτό κάνουμε εμείς σε καθημερινή βάση 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε τον ανθρώπινο πόνο, ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν μέσω θαλάσσης και αν δεν τους σώσουμε εμείς θα βρουν σίγουρα θάνατο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δέχτηκα με ενθουσιασμό αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη δραστηριότητα τη Ιταλικής ακτοφυλακή στην περιοχή μας. Θα κάνω μια σύντομη ανάλυση και θα σα δώσω πληροφορίες για το πώς ακριβώς επιχειρούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Η μετανάστευση, η θαλάσσια προς την Ευρώπη αφορά ιδιαίτερα την Ιταλία. Ξεκίνησε το 1991 αυτό το φαινόμενο με τη μετανάστευση από την Αλβανία και απέκτησε συστηματικό χαρακτήρα με τις ροές μετά από τις σειράξεις στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή οδηγώντας τον συντονισμό διάσωσης πάνω από 600.000 600 άτομα. και έχουμε σώσει πάνω από 324.000 άτομα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε η Δήμαρχος Νικολίνη που μίλησε προηγουμένως που είπε από τις 3 του Οκτώβρη μέχρι σήμερα τα τρία τελευταία χρόνια έχουν πεθάνει 11.500 άνθρωποι. Αν δεν υπήρχε η οργάνωσή μας και όταν μιλάω για οργάνωσή μας μιλάω για χώρες βέβαια στο σύνολό τους, για την Ιταλία συγκεκριμένα και χάρη στις, ε, στην βοήθεια που έχουμε στην θάλασσα, γιατί όλοι βοηθούν στη διάθεση όσο εκεί. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο σώσαμε 500.000 άτομα. Θα ήθελα λοιπόν να το τονίσω αυτό, δηλαδή να δούμε τη σημασία που έχει η παρουσία η δικιά μας στη θάλασσα και ο συντονισμός τόσων δημοσίων αρχών και τόσων ατόμων για την διάσωση. Ανέκαθε συμμετείχε λοιπόν η ακτοφυλακή Ιταλική στην διάσωση σε σχέση με 7 διαφορετικές μεταναστευτικές ροές. Προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, η φυσική ροή δηλαδή από την Αφρική πέρα προς την Ιταλία, από την Ανατολική Μεσόγειο, Αίγυπτος, Τουρκία και από την ε, Αδριατική και το Ιόνιο, Ελλάδα και Αλβανία. Η κάθε ροή έχει δικές της ιδιαιτερότητες όσον αφορά την διοργάνωση, την εγκληματική, την τυπολογία, τις εθνικότητες και τους μετανάστες που εμπλέκονται. Οι κύριες ροές προέρχονται από την Λιβύη, 89% των ατόμων που έχουν διασωθεί, και 10% από τις ακτές της Αιγύπτου. Αν σκέφτεται κανείς λοιπόν γιατί καθημερινά συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης η ακτοφυλακή. Ο κίνδυνος μεγάλων απολειών ανθρώπινων ζώων είναι πολύ ψηλό. Ο κύριος λόγος, η κύριοι είναι το ότι καταρχάς έχουμε σκάφη τα οποία είναι χειροποίητα και δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό. Η έλλειψη επίσης εξειδικευμένου προσωπικού η... ο μεγάλος αριθμός ε, ατόμων στα σκάφη αυτά που θέτει τη ζωή σε κίνδυνο, η έλλειψη μέσων διάσωσης και η παρουσία σε αυτά τα σκάφη περιπτώσεων όπως άτομα με προβλήματα αμαία, έγκυες γυναίκες κλπ. Να σας πω ότι μόνο χθες σώσαμε 1.004 άτομα και αυτά τα άτομα οδηγήθηκαν στην ε, Κατάνια, αλλά έφτασαν 1.007 επειδή γέννησαν τρεις γυναίκες. Η Ιταλική Ακτοφυλακή επίσης δρά εκτός των ορίων δικαιοδευσίας της προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες ότι το πρώτο κέντρο διάσωσης το οποίο λαμβάνει γνώση του κινδύνου σε μια περιοχή εκτός της ε, περιοχής Search and Rescue θα πρέπει να στείλει αμέσως σήμα και μέχρι να αναλάβει την ευθύνη της διάσωσης το κέντρο αυτό θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό της διάσωσης. Τώρα τι γίνεται, από το 11 και μετά η Λιβύη με την άνοιξη του εμφυλίου δεν έχει πια τη δυνατότητα να διασφαλίσει τον ε, συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης. Οπότε στάθηκε απαραίτητο να εμπλακεί όλο και περισσότερο η Ιταλική Ακτοφυλακή που χρειάστηκε να παρενέβει πέραν των υδάτων δικαιοδοσίας της. Επειδή η έκκληση διάσωσης ε, προέρχεται από άλλο κέντρο. Φτάνουν λοιπόν στην Ιταλία αυτέ οι εκκλήσει για διάσωση. Οπότε η Ιταλία θα πρέπει να διασφαλίσει την παρέμβαση διάσωση, επειδή η Λιβύη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη. Αναβάλλει λοιπόν το συντονισμό η Ιταλική ακτοφυλακή όλων των πτυχών τη διάσωση. Εδώ και καιρό καθημερινά συμμετέχουν και στρατιωτικέ δυνάμει υπό το τρίτονα τη Ευρωπαϊκή ε, δυνάμει. Έχουμε και τις μονάδες υποεθνικό έλεγχο, ναυτικό, ε, αστυνομία, λιμενικό και συμμετέχουν ακόμα και αλληλείς, όπως και σκάφη μη κυβερνικών οργανώσεων που μας βοηθούν πολύ. Οι ΜΚΟ πραγματικά συμβάλλουν τα μέγιστα στη διάσωση. Ελήψη λοιπόν εταίρων στο νότο της Μεσογείου η Ιταλική ακτοφυλακή είναι η μόνη αρχή de facto διάσωσης που είναι παρούσα σε μία έκταση 1,2 τετραγωνικών, 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή η μισή Μεσόγειος. Η ροή από το 2014 συνεχίζεται και αυξάνεται. Το 2016 έχουμε παρόμοια στοιχεία με πέρσι, δηλαδή αφήξει γύρω σε 150.000 μεσοθαλάσσιες. Τις τελευταίε εβδομάδες ήδη έχουμε φτάσει στι 145.000, οπότε υποθέτω ότι δυστυχώς αυτό το στοιχείο θα αυξηθεί. Τροφοδοτείται κυρίω αυτή η ροή από αφρικανικές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και οι υπόλοιπε χώρε ε, και οι υπόλοιπε ανικότητε είναι κυρίω από Νιγηρία. Χρησιμοποιούνται κυρίω σκάφη ξύλινα και έχουμε αύξηση και των σκαφών που έχουν διασωθεί φέτος ας πούμε κατά 10%. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται 12 μέτρα με 120 άτομα περίπου λόγω ακριβώς της τεχνικής που χρησιμοποιείται τα σκάφη αυτά έχουν δυνατότητα πλεύσης για ελάχιστες, ελάχιστες ώρες και θα πρέπει να διατρέξουν 35 ναυτικά μίλια. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η αναχώρηση μέσων που χρησιμοποιούν οι μετανάστες, τα οποία έχουν πλημμυρίσει και που το 16 ας πούμε, καταγράψαν 58 τέτοιες αναχωρήσεις. Χρειάστηκε να κάνουμε παρεμβάσει 58 τέτοια σκάφη τα οποία είχαν, φύγει, είχαν ξεκινήσει την ίδια μέρα. Χρησιμοποίησαν δηλαδή μετανάστες οτιδήποτε έπλεε και σώσαμε 7.000 άτομα εκείνη την μέρα μόνο. Εξάλλου η συστηματική καταστροφή αυτών των ε, σκαφών μείωσε δραστικά τον αριθμό τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο να παρενέβουμε στα αίτια αυτής της ροής. Για τη Συρία τώρα. Βλέπουμε να υπάρχει κάποια μείωση εδώ και κάποιους μήνες από τη στιγμή που έχουμε τη συμφωνία με την Τουρκία. Οι Σύριοι δεν προβλέπουν πια την ε, μετάβαση από τη Μεσόγειο παρά μόνο σε πολύ χαμηλούς αριθμούς. Και οι ίδιοι έχουν δυνατότητα οικονομική μεγαλύτερη, μπορούν να πληρώσουν τους διακινητές. Και επειδή ακριβώς υποχώρησε αυτή η ροή. Έχουμε μείωση των αριθμών. Πού οδήγησε όμως ε, αυτό. Αυξήθηκε το κόστος για τις υπόλοιπες ροές. Αυξήθηκε το κόστος ας πούμε των, ε, των καυσίμων και οι διακινητές έχουν γίνει πιο αυστηροί, πιο ληστρικοί σε σχέση με τους μετανάστες. Και χθε να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα φουσκωτό τελείως τυχαία λίγο έξω από τα λιβικά ειδικά τελείως τυχαία εντοπίστηκε από μια μονάδα μας και βέβαια διασώστηκε εμείς δεν είχαμε καμία επικοινωνία σε σχέση με αυτό το φουσκωτό και την αγχώρησή του γιατί συνήθως ε, έχουμε ένα στίγμα μέσω δορυφόρου για κάθε σκάφος για να εξοικονομήσουν λοιπόν χρήματα οι διακινητέ, δεν δίνουν δυνατότητα σε αυτά τα άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλε δυσκολίε να δώσουν κάποιο στίγμα. Δεν τους δίνει λοιπόν ούτε καν τη δυνατότητα να τηλεφωνήσουν στις, ε, στους ε, διασώστες. Η κεντρική λοιπόν Μεσόγειος είναι ένα θέατρο που περιέχει μεγάλες αποστάσεις 150 χιλιόμετρα η απόσταση, ας πούμε, Βρυξέλλες, ε, Παρίσι, μέχρι να φτάσει και στη Λαπεντούσα. Πάντως στη Λαπεντούσα έχει επιδείξει η τοπική κοινότητα μεγάλη αλληλεγγύη και έχει υποδεχθεί θερμά τους μετανάστες. Τώρα για τα εναέρια μέσα θα πρέπει να βρεθούν μέσα με μεγάλη αυτονομία ή εναλλακτικά ελικόπτερα. Η κεντρική Μεσογείο χρειάζεται λοιπόν πιο περίπλοκα και πιο ακριβά μέσα διάσωση σε σχέση με τα μέσα διάσωση που χρησιμοποιούνται σε άλλε θάλασσε, ε, όπω το Αιγαίο α πούμε. Ξέρουμε τι γίνεται στα ελληνικά νησιά, Σάμο, Κο, όπου οι αποστάσει είναι πολύ μικρέ 1-1,5 μίλι. υπάρχουν διαφορετικοί κινδυνοί εκεί, ίσως οι άνεμοι κτλ. Όμως σίγουρα δεν έχουμε να κάνουμε 250 χιλιόμετρα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Οι μεγάλοι αριθμοί λοιπόν που αντιμετωπίζουμε απαιτούν καταρχάς τη συνεχή παρουσία ειδικευμένων ε, δυνάμεων και την ε, αρρωγή από σκάφη έτοιμα ώστε να έχουμε την κατάλληλη μεταφορά των ατόμων αυτών στη στεριά. Και εδώ να σας δώσω πάλι ένα πρακτικό παράδειγμα. Έχουμε τα σκάφη του ναυτικού που όμως είναι εκεί για συγκεκριμένου λόγους. Παρεμβαίνουν επειδή ακριβώς βεβαίως προβλέπει διά, η διάσωση. Όμως εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στην δικιά του την αποστολή. Και υπάρχουν και άλλες μονάδες που έρχονται κοντά σε αυτά τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ώστε να γίνει μετά η αποβίβαση των ατόμων αυτών στη στεριά. Και αυτή λοιπόν η δραστηριότητα καθημερινά συντονίζεται από το επιχειρησιακό κέντρο τη ακτοφυλακή. Εδώ επίση πρέπει να προσθέσουμε το γεγονό ότι δεν μπορούμε πάντοτε να διασφαλίσουμε την μεταφορά των μεταναστών στα hot spot γιατί μπορεί να υπάρξουν ε, απρόβλεπτες ανάγκες ε, διάσωσης. Οι ναυτικές λοιπόν μονάδες ως βοηθητικό μέσο θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο ώστε να γίνει σωστός καταμερισμός ακριβώς της διασωστικής προσπάθειας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω μόνο ότι Πέρσι και, ε, συγγνώμη, χθες και προχθές διασώσαμε 10.600 άτομα. Αυτά όμως τα 10.600 άτομα δεν μπορούν να μεταφερθούν αποκλειστικά στα hot spots στη Στεριά, στο Ποτσάλο, στην ε, Λαμπεντούζα, στο Τράπανη και αλλού. Είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να γίνει μια κατανομή έτσι πιο ευρεία στην επικράτεια. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε 10.600 άτομα σε ελάχιστα σημεία, γιατί σήμερα μιλάμε ας πούμε για 1.000 άτομα χίλια άτομα, το οποίο πιο εύκολο το διαχειρίζεται από 10.600. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και, ο, και η ανάγκη και, ο, και επιβάλλεται να γίνει μια πιο ευρεία κατανομή αυτών των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε όλοι ότι η Ιταλία συμβάλλει καθοριστικά, γιατί συμμετέχουν οι περιφέρειες, οι, οι τοπικές αρχές, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι ΜΚΟ, όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη διάθρωση, πέρα βέβαια από την δικαιοσύνη. Η Ιταλική ακτοφυλακή λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στο συντονισμό βέβαια και σε αυτές τις δράσεις, αλλά χάρη και στη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές επέτρεψε την ε, καταπολέμηση της έναρξης αυτής της ροής. Έχουν ήδη συλληφθεί διακίνητες αρκετοί τα δύο τελευταία χρόνια μετά από εντελεχείς έρευνες και Παρενέβη επίση η Ιταλική ακτοφυλακή σε δίκτυα διακινητών με πάνω από 26 συλλήψεις. Εν απουσία λοιπόν ανθρωπιστικών διαδρόμων ή άλλων λύσεων που θα αποτρέπουν την αναχώρηση των μεταναστών, μόνο η θαλάσσια διάσωση αποτελεί τον τρόπο αποφυγής απώλειας ανθρωπίνων ζώων. Θα πρέπει λοιπόν όποιο προσπαθεί να έρθει στην Ευρώπη να εντοπίζεται και να είμαστε σε θέση να τρέξουμε στην πηγή της εκμετάλλευσης. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε την ασφάλεια των, των θαλάσσιων συνόρων μας και την ανάγκη διασφάλισης της αξίας ανθρώπινης ζωής και της διάσωσής της. Όταν εμείς μεταφέρουμε στα σκάφη και στις μικρές και στις μεγάλες ομάδες τους μετανάστες αυτούς. Εδώ και 25 χρόνια το κάνουμε αυτό. Το προσωπικό μας έχει αποκτήσει πολιτή εμπειρία και μπορεί να εντοπίσει κιόλα τους διακινητές. Σε ένα λοιπόν συγκεκριμένο περιβάλλον ή πλαίσιο του σκάφους είναι εύκολο από εκεί ήδη να, να κατανοήσουμε ποιος είναι ο διακινητής. Γι' αυτό ακριβώ λοιπόν και η αστυνομική δραστηριότητα ξεκινάει από τη θάλασσα και μετά φτάνουμε στη, στη, στεριά, φτάνουμε αυτά, τα άτομα αυτά παραδίδονται στι αστυνομικέ δυνάμεις και μετά συνεχίζεται η συνήθεια διαδικασία. Γιατί σα το λέω αυτό. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, εδώ και καιρό λέμε, γιατί δεν δημιουργούμε κινητά hot spot, δηλαδή γιατί δεν δημιουργούμε ας πούμε hot spot με σκάφη, με πλατφόρμες οργανωμένες ώστε να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες σε αυτά τα σκάφη ώστε να γίνονται και εκεί όλες οι αστυνομικές ε, ενέργειες σε ένα κλειστό περιβάλλον. Θα ήταν πολύ πιο απλό ώστε με, στη συνέχεια με τη σειρά τους τα σκάφη αυτά να είναι σε θέση να κάνουν μια κατανομή πιο ε, ισοβαρή στα διάφορα μέρη της χώρας. Όπως είδατε στο φιλμ στην αρχή, έχουμε μια πρωτοβουλία πρεσβευτών, 38 πρεσβευτών από αφρικανικές χώρες που στην Ρώμη έδωσαν μια αναμνηστική, αναμνηστική πλακέτα ως χειρονομία αναγνώρισης της συμβολή της στις ε, ενέργειες διάσωσης Κανένας άλλος παγκόσμιος οργανισμός δεν έχει διασώσει τόσες ανθρώπινες ζωές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με τέτοια συχνότητα ώστε να έχει μετατρέψει δυστυχώς τη διάσωση σε καθημερινό συμβάν. Πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με το capacity building ώστε να είναι σε θέση η Ιταλική ακτοφυλακή να βοηθήσει και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αρχές, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ακτοφυλακές στην κατάρτισή τους για τις σωστές επιχειρησιακέ επιχειρησιακές αυτού του είδους. Θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων και θα πρέπει οι ευρωπαϊκές αρχές να συνεργαστούν γι' αυτό. Η συνεργασία διέρχεται βέβαια και από την προώθηση των πρωτοβουλειών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για, τις, ε, για τη λειτουργία της ίδιας της ε, ακτοφυλακής. Αυτό το φόρουμ είναι ένας άξιος και χρήσιμο συνομιλητή, επειδή ακριβώ συγκεντρώνει όλου του φορεί που εμπλέκονται στι δράσει των ακτοφυλακών. Αυτή η ενέργεια λοιπόν και η ανάπτυξη πρέπει να έχει προτεραιότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ιταλική λοιπόν ακτοφυλακή με τη βοήθεια της Κομισιόν ξεκίνησε ένα φόρουμ που τον περασμένο Ιούλη στην ε, Νάπολη είδε και τεράστια, είχε και τεράστια συμμετοχή από ακτοφυλακές της, Ευρώπη, της, ε, της Μεσογείου, την Ισία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Τουρκία. Αποφάσιστηκε λοιπόν να ξεκινήσουν κάποιες δραστηριότητε συνεργασίας σε επίπεδο κατάρτισης, ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε καλύτερα η δέσμευση της Ιταλικής ακτοφυλακής είναι καθημερινή και συνίσταται σε ανθρωπιστικές βοήθειες για την διασφάλιση του απότερου αγαθού της ανθρωπινής ζωής. Τώρα όμως προστίθεται και βέβαια και η διασφάλιση του θαλασσίου περιβάλλοντος, η επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας ώστε να έχουμε όλο και πιο ασφαλή πλεύση. Επίσης στρέφεται και προς το μέλλον μέσω του capacity building και να σα πω για το λεφτό αυτό σημείο ότι με περηφάνεια δέχτηκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόκληση για την συγκρότηση του Λιβικού Κέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης. Αυτό αποτελεί και μια μεγάλη αναγνώριση της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Ιταλική Ακτιοφυλακή στον τομέα της διάσωσης. Έχουμε και το πρόγραμμα Σοφία για την κατάρτιση της ε, λιβικής ακτοφυλακής. Και θα ήθελα τώρα να τελειώσω λέγοντας τα εξής. Η ακτοφυλακή καθημερινά κάνει διασώσεις, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις παράνομες ροές και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την υποδοχή των ατόμων που έχουν φύγει, ότι, που είναι πρόσφυγες, ως ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα. Τα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα λοιπόν θα πρέπει να ανατεθεί το έργο της διασφάλισης της εφαρμογής αυτής της αρχής που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα. Έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά μέρη, μακριά από την πατρίδα τους, δεν μιλούν τις γλώσσες και είναι σε κατάσταση, είναι ευάλωτη. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό που είχε πει ο πρόεδρος Ρούσβελτ σε μια σημαντική ομιλία του 41 σε σχέση με τις τέσσερις ελευθερίες ότι έχουμε ελευθερία έκφρασης, ελευθερία πίστης, ελευθερία από, την, από το φόβο και από την ανάγκη. Στο Κογκρέσο το Αμερικανικό με λίγα λόγια λοιπόν αλλά πολύ αποτελεσματικά είπε ο Ρούσβελτ ότι δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικές ελευθερίες ατομικές και συλλογικές αν συνεχίζει να κυβερνάει ο φόβος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Θα πρέπει να πούμε ότι ο δρόμος του διαλόγου περνάει από την Ευρώπη η οποία διδάσκει ότι η αμοιβαιότητα και η βοήθεια προς τους μετανάστες πρέπει να επεκτείνεται και στους πολιτισμούς τους. Το φαινόμενο αυτό δεν ε, δέχεται μια μοναδική απάντηση. Θα πρέπει να πάμε στα αίτια, στα βαθιά αίτια αυτού του φαινομένου. Πάντως θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι εσάς για την πρόσκληση και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πάντοτε θα υπάρχει στο πλάι σας η του Ακτοφυλακή. Ευχαριστώ. Vielen Dank, σας ευχαριστώ πολύ, και Μελώνε. Σα ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή, εξαιρετικά διαφωτιστική. Το επαναλαμβάνω, επειδή εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, είμαι πολίτη και πράγματι... Ακούσαμε αυτά που μόλις είπατε και νομίζω ότι... Ε, Κύριε Υποπλήρχε, θα ήσασταν πολύ καλός ευρωβουλευτής. Ε, πράγματι έχετε το δώρο του λόγου. Ακούσαμε τώρα το πολεμικό ναυτικό ε, της Ιταλίας. Ε, τώρα περνάμε στην επιχείρηση Σοφία που αποτελεί μέρος της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Κύριε Υποπλήρχε Κρεδεντίνο, σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνεται τη δυνατότητα να παρουσιάσω την επιχείρηση Σοφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η επιχείρηση μάλιστα έλαβε το όνομά της από ένα πλοίο του, ε, Ιταλικού, ε, της Ιταλικής Ακτοφυλακής. Και με αυτόν τον τρόπο ε, μιας και η επιχείρηση ε, περιστρέφεται γύρω από τις δραστηριότητες τις οποίες εμείς έτσι και αναπτύσσαμε εδώ και πολύ καιρό θα ονομαζόταν ε, με αυτόν τον τρόπο. Σοφία. Το 2015 είχαμε την μεγαλύτερη καταστροφή, το μεγαλύτερο ναυάγιο που είχαμε ποτέ δει μέχρι τότε στη Μεσόγειο με 800 νεκρούς και ε, ε, μετά από αυτό το περιστατικό κινητοποιήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων εξωτερικών και ε, δημιούργησε το σχετικό πρόγραμμα δράσης για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης με μια ολιστική προσέγγιση και με στόχο να καταπολεμηθούν οι γενουσιεργές αιτίες τα βαθύτατα αίτια που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους να καταλήξουν τις αιστείες τους. Αναγνωρίστηκε λοιπόν η ανάγκη να εργαστούμε με τέτοια προσέγγιση, με ε, συνολική προσέγγιση. Ε, η εντολή λοιπόν που μας δόθηκε είναι εξαιρετικά σαφής. Στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων στη Μετσόγειο δεν ε, συμπεριλαμβάνονται στην ε, εντολή μας οι ε, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά φυσικά, όπως είπε και ο συνάδελφος υπονάβαρχος πριν, είμαστε άνθρωποι της θάλασσας, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αφήσουμε έναν άνθρωπο να πνίγει. Είναι ζήτημα ηθικό για εμάς. Επομένως πάντοτε, οποτεδήποτε κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει στη θάλασσα, φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον διασώσουμε. Είμαστε ε, η μόνη επιχείρηση στην οποία συμμετέχει η αεροπορία και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε πότε ξεκινάει ένα πλοίο από τη Λιβύη και ε, ενημερώνουμε πάντα και συνεργαζόμαστε και με την ύπατη ε, εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Σήμερα 25 φορες μέλη συμβάλλουν με προσωπικό ή σκάφη ή με συγχρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχής χωρομελών σε ευρωπαϊκή επιχείρηση, όπως ρεκόρ ήταν και ο σύντομος χρόνος έναρξης της επιχείρησης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι χώρες μέλη είχαν τη βούληση να θετήσουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση ενό ορού προβλήματο. Η επιχείρηση είχε τέσσερι φάσει. Η πρώτη ήταν η συλλογή πληροφοριών και η παρουσία τη δύναμη στην θάλασσα. Τώρα βρισκόμαστε στην φάση όπου προσεγγίζουμε τα ύδατα της Λιβύης για να καταπολεμήσουμε τους διακινητές στην ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε την 2240 του ΟΗΕ ως ψήφισμα που μας επιτρέπει αυτή η δραστηριότητα σε διεθνή ύδατα. Η επόμενη φάση είναι να πάμε στα χωρικά υδατά της Λιβύης, αλλά χρειάζεται πρόσκληση της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης και νέο ψήφισμα του ΟΗΕ. Και βεβαίως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πώς θα λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, δηλαδή τους διακινητές που θα θέλαμε να συλληφθούν εντός χωρικών υδάτων Λιβύης. Πάντως όποιος συλλαμβάνεται σε διεθνή ύδατα οδηγείται στην Ιταλία. Αυτό το κάνουμε από την αρχή. Και αυτές είναι και οι οδηγίες που είχαμε από την αρχή της επιχείρησης. Η άλλη απόφαση είναι η αρχή της μη απόθεσης. Κανένας λοιπόν μετανάστης δεν μπορεί να οδηγηθεί σε τρίτες χώρες. Αυτό όμως το μοντέλο το να οδηγηθούν όλοι και διακινητές και μετανάστες στην Ιταλία αυτό λοιπόν το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα χωρικά δετά της Λιβύης δηλαδή αν συλλάβουμε διακινητές σε εθνικά ύδατα της Λιβύης θα πρέπει να δώσουμε στις λιβικές αρχές τους λιφθέντες κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν υπάρχει συμφωνία οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αφήσουμε ελεύθερους κάτι το οποίο ακυρώνει την επιχείρηση πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πριν πάμε στα χωρικά ύδατα της Λιβύης μπορεί να λυθεί αυτό μόνο μέσω διμερούς συμφωνίας χώρας μέλους Λιβύης ώστε μετά να δικαστούν στην χώρα μέλος αυτοί οι διακινητές. Σήμερα δικάζουμε στην Ιταλία αυτούς που βρίσκουμε στα διεθνή ύδατα. Αν λοιπόν η Ιταλία συνάψει διμερή σχέση με τη Λιβύα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Άλλη δυνατότητα είναι η Συμφωνία Λιβύης Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι το οποίο θα ήταν καλός μακροπρόθεσμη λύση. Γιατί πολύ συχνά αυτοί οι διακινητές βρίσκονται σε απάνθρωπες συνθήκες στις λιβικές φυλακές. Μέχρι λοιπόν να λύσουμε το νομικό ζήτημα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την επιχείρηση. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε στα χωρικά εδατά της Λιβύης. Για να λύσουμε αυτή λοιπόν την, κατάσταση, να βρούμε μια λύση, κάνουμε το εξής. μέχρι την συμφωνία με την Τουρκία το 90% έμπαιναν μέσω Βαλκανίων. Μόνο το 10% Λιβύη η Ιταλία. Από τις 4 το Απρίλη από την θέση ισχύ της συμφωνίας το 90% έρχεται από την Ιταλία. Οι αριθμοί σε σχέση με πέρσι δεν έχουν αλλάξει πολύ και από τη Λιβύη και την Αίγυπτο καταφθάνουν άτομα από την υποσαχάρια Αφρική. Φέτος είχαμε πάνω από 3.000 νεκρούς μετανάστες που ήρθαν από τη Λιβύη. Η πλειοψηφία τους πεθαίνει είτε στα χωρικά ύδατα της Λιβύης πολύ κοντά. Και αυτό επειδή εμείς δεν είμαστε σε θέση να παρενεύουμε, επειδή είμαστε πολύ μακριά, δεν έχουμε την νομική δυνατότητα. Με το Σοφία εμείς θέλουμε να καλύψουμε όλη την Λιβική επικράτεια, όπου υπάρχουν πολλές δροές και άλλες επιχειρήσεις, ο Τρίτονας, η, η Σίγουρη Θάλασσα, η Ασφαλής Θάλασσα Ιταλική, και άλλες επιχειρήσεις. Έχουμε και ΜΚΟ και έχουμε και το ΝΑΤΟ το οποίο βρίσκεται να άξονα Ανατολή δράσεις και παρεμβάσεις. Όλα αυτά μετά συντονίζονται από την τελική ακτοφυλακή όσον αφορά τη διάσωση. Ακτοφυλακή η οποία ευτυχώ είναι σε θέση να παρενέβει και να δεσώσει πολλές ζωές. Έχουμε τρία αεροσκάφη περιπολικά, έχουμε και ελικόπτερα και είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τέτοια θαλάσσια δύναμη στη Μεσόγειο. Και αυτό βεβαίω συμβάλλει στην ασφάλεια του Μαρενόστρομ, στρατηγική σημασία βέβαια, όχι μόνο για την Ιταλία αλλά για όλε τι μεσογειακέ χώρε. Πρόσφατα είχαμε άλλες δύο αρμοδιότητες που προστίθεται στην αρχική εντολή για την καταπολέμηση των διακινητών και που χρειάζονται για την επίτευξη της επιχείρησης. Έχουμε το training και το capacity building της λιβικής ακτοφυλακής σε αυτή την αρχική φάση. Δεν έχουν ε, δυνατότητα ένοπλης αντίδρασης, αλλά βρισκόμαστε στην πρώτη φάση κατάρτισης. Για την κατάρτιση τώρα συγκεκριμένα της Λιβικής Ακτοφυλακής, να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε κατά τα τέλη του τρέχοντα μήνα τις ενεργειές μας. Ήδη έχουν έρθει οι πρώτοι 80 Λίβοι. Η εκπαίδευση γίνεται σε δύο σκάφη, ένα Ιταλικό και ένα Ολλανδικό. Στις 24 του Οκτώβρη προβλέπεται η άφηξή τους. 14 εβδομάδε λοιπόν σε διεθνή ύδατα θα γίνει εκπαίδευση αυτών των Λιβύων ακτοφυλάκων. Και προβλέπουμε να φτάσουμε σε 500 ή 600 ώστε το Μάρτι του χρόνου να έχουμε άτομα τα οποία θα έχουν καταρτιστεί για όλες τις δραστηριότητε της ε, ακτοφυλακής. Έχουμε και σκάφη τα οποία θα θέλαμε να δώσουμε. Εμείς δεν είμαστε στρατιωτική ακτοφυλακή, εμείς υπαγόμαστε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά για την άνοιξη του 17 θα θέλαμε η Λιβική ακτοφυλακή να είναι σε θέση να κάνει περιπόλους και να μπορείς να καταπολεμήσει όχι μόνο τη διακίνηση, διακίνηση όχι μόνο μεταναστών, αλλά και όπλων, ναρκωτικών κτλ. Αλλά και να κάνει και τις διασώσεις. Αφού λύσουμε βέβαια και το θέμα το νομικό, γιατί όπως σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχει να φαινόνται ελεύθεροι. Και επίσης βέβαια για να μην έχουμε και τόσους νεκρούς όπως είχαμε, όσους είχαμε φέτος και όπως είχαμε φέτος στα λιβικά χωρικά ύδατα. Δεύτερο σημείο. Εμπάρκο όπλων για τη Λιβύη. Είχαμε πρόσφατα την 2292, το 2292 ψήφισμα του ΟΗΕ που μας επιτρέπει ακριβώ να ελέξουμε εμπορικά πλοία για τα οποία υπάρχουν υποψίες για παράνομο εμπόριο όπλων. Αυτή η δραστηριότητα είναι αρκετά δύσκολη. Και οδηγεί σε επικίνδυνε καταστάσει όταν ακριβώ όντω μεταφέρονται όπλα και υπάρχουν και τρομοκράτε στα πλοία που δεν θέλουν να σταματήσουν. Δεν σταματάμε όταν δεν σταματάμε όταν ελέγχουμε. Αυτές είναι οι δραστηριότητες λοιπόν που έχουμε και άλλη μια σημαντική δραστηριότητα την οποία διευθύνω εγώ είναι οι επαφές με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς επαφές σε επίπεδο υπουργών, γενικών γραμματείων υπουργείων, ΟΗΕ, ιδιαίτερα την υπατιαρμοστία για τους πρόσφυγες Θα μας βοηθήσει λοιπόν είπατε η αρμοστία και στην εκπαίδευση ακριβώς της Λιβικής Ακτοφυλακής και μας βοηθάει επίσης και σε άλλα θέματα θέματα φύλου την προστασία των παιδιών κλπ. Έχουμε στενή σχέση και επαφή και η παρουσία Ιταλών αξιωματούχων στην πατερμοστία μας διευκολύνει Έχουμε επίση και στην συνεργασία με την Frontex, με την οποία έχουμε επίσημη συμφωνία. Έχουμε ανταλλαγή προσωπικού, ανταλλαγή αξιωματικών και προσπαθούμε γενικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της διακίνησης μαζί με άλλες διεθνείς αρχές όπως Europol, Eurojust, τα Ηνωμένα Έθνη και διάφορες άλλες ε, υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών μελών και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να συγκροτούμε το παζλ αυτό το μοσαϊκό. Αντιμετωπίζουμε επίση και φαινόμενα πειρατείας, αλλά πολύ λιγότερο. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στον ΟΗΕ και είχαμε πολλές επαφές με την υπάτη αρμοστία. Πάντως η επιχείρησή μας είναι γνωστή, τη γνωρίζουν όλοι και πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με την περιφερειακή μας δράση και παρουσία όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Και έχουμε αυτό το μηχανισμό αναφόρουμ όπου έχουμε όλες τις οργανώσεις των χωρών που εμπλέκονται στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Το Νοέμβρη πέρσι είχαμε την τελευταία συνάντηση, 74 οργανισμοί συμμετείχαν ΜΚΟ, ναυτιλιακές εταιρείες, ΟΗΕ, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Είχαμε και εννέα ομάδες εργασίας με διαφορική θεματολογία για να προσπαθήσουμε έτσι όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Συνοψίζοντας να σας πω ότι το Σοφία είναι ακριβώς η υλοποίηση τη βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εντοπίση αυτού του προβλήματο. Βρισκόμαστε βέβαια στην αρχή, βρισκόμαστε στη φάση κατανόηση αυτού του φαινομένου. Προσπαθούμε να δούμε πώ ε, επιχειρούν οι διακινητέ. Θα πάω και στην Αντίσα Μπέμπα σύντομα. Θα συναντήσω και προσώπους της ε, Αραβική Ένωση ε, στη ΣΥΠΑ. Και πάντως αυτά που κάνουμε έχουν αποτέλεσμα γιατί οι διακινητές υποχρεώνονται να παραμείνουν στα λιβικά χωρικά υδατά μετά από τις δράσεις μας και ξέρουν ότι αν βγουν από τα χωρικά υδατά της Λιβύης θα συλληφθούν και θα καταστρέψουμε το σκάφος που θα μεταφέρουν. Έχουμε διασώσει λοιπόν πάνω από 7.000 ζωές και έχουμε παραδώσει στην Ιταλική δικαιοσύνη 89 διακινητές και έχουμε εξοδοτηρώσει πάνω από 300 σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν διακινητές για αυτό το είδος απάνθρωπης διακίνησης. Και έχουμε λέξει 52 εμπορικά σκάφη που θα μπορούσαν να μεταφέρουν παράνομα όπλα στην Λιβύη. Αυτά πρόεδρε από Είμαι στη διάσταση να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κρεντεντίνο. Η ώρα πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ομιλίες σας. Ευχαριστώ την Τζούσα Νικολίνη. Προτείνω να συμφωνήσουμε όλα τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ε, να τα αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Και ο πρόεδρος παρακαλεί τους διερμηνείς ε, να παραμείνουν λίγα λεπτά ακόμα, διότι έχουν ζητήσει κάποιοι το λόγο. Δύο λεπτά μας μένουν ακόμα. Να δούμε πόσο θα προχωρήσουμε. Έχουμε περιορισμένο χρόνο λόγω διερμηνίας. Κατανοητό ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς ε, διερμηνία πάρα πολύ ώρα. Ε, προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε κατευθείαν ε, στους ομιλητές. Η κυρία Τσουνίση κατόπιν hatte Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα τους τέσσερις συναδέρφους. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω Αντί για 10 να μιλήσω ένα λεπτό. Χαιρετίζω την Δήμαρχο Κολίνη που γνωρίζω εδώ και καιρό και χαιρετίζω ιδιαίτερα όλους τους πολίτες της Λαμπεντούζα καθώς και τους Ναβάρχους και την Ιταλική Ακτοφυλακή. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας γιατί ως Σικελή και Ιταλίδα γνωρίζω την προσπάθεια των αρχών και των απλών πολιτών για την υποδοχή των μεταναστών. Θα είμαι σύντομη. Στην Ευρωβουλή ασχολούμαι με τα θέματα των ανηλίκων, για του οποίους έχουμε μια ομάδα εξειδικευμένη και που αποτελούν την πιο ευάλωτη πτυχή αυτού του φαινομένου. Και στα hot spot προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί δυστυχώς ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων και για να συντομεύσω να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση. Τι γίνεται και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Ο αντιπρόεδρος Τιμέρμαντς πήγε στην Σικελία αρχές Σεπτέμβρη και ο ίδιος είπε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα. Λαμβάνοντας υπόψη και τη δουλειά που έχει στη Σικελία, με την παροχή αρρωγής, ψυχολογικής, ιατρικής κλπ. Στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ των αρχών μας. Οπότε ρωτάω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και εμείς ως Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να στηρίξουμε ακριβώς το πιο αδύναμο κομμάτι, το πιο αδύναμο τμήμα των μεταναστών προχώρησης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία Τσουφρίδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια προς την ακτοφυλακή μας και για την συνάντηση αυτή που διοργανώσαμε. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο συγγνώμη, τη Δήμαρχο Νικολίνη που μίλησε σκληρά αλλά είπε την αλήθεια και είπε ότι είναι καταθλιπτικό αυτό που βλέπει κανείς στην Λαμπεντούζα και είναι ακόμα περισσότερο αν δούμε την αδράνεια και την αδιαφορία κάποιων μπροστά σε εικόνες που είναι καθημερινή πραγματικότητα στην απαιτούσα και αλλού. Εγώ λοιπόν ρωτάω προκλητικά. Μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε αυτές τις εικόνες και μήπως θα έπρεπε να ξανακάνουμε τέτοιες συναντήσεις ώστε αυτή η πραγματικότητα να γίνει περισσότερο γνωστή. Γι' αυτό να καλέσουμε τον κύριο Νόρμπαν, τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Αφού λοιπόν έχει τοποθετηθεί επανειλημμένο το Κοινοβούλιο, αφού επιτέλου επιτέλους, η Κομισιόν μα έδωσε ένα σχέδιο επανεγκατάσταση, το οποίο όμω βρίσκεται σε αδράνεια, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το Συμβούλιο συνεχίζει να καθυστερεί. Γιατί είπε η Δήμαρχος και είπε σωστά τι προάλλες ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μόνο λόγια τη στιγμή που έχουμε 11.000 νεκρούς. Ρωτάω λοιπόν εγώ και εμείς εδώ συνάδελφοι αναρωτιόμαστε πού διακρίνονται οι θεσμοί. Γιατί το κοινοβούλιο είναι συμπαγές αυτό. Η Κομισιόν είπε ότι έχουμε δίκιο. Έχει έρθει όμω τώρα η στιγμή επιτέλους να αναλάβουμε μια ισχυρή δράση ώστε επιτέλους το Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις και να μην υπάρχουν πια χώρες μέλη οι οποίες ενώ ωφελούνται από την Ευρώπη παραβλέπουν και παρακάμπτουν τους κανόνες που η ίδια η Ευρώπη ε, θέλει να εφαρμόσει. Ευχαριστώ κύριο Σπανιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι... Ε, μας συγκίνησαν. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μας δείξατε και μας ανησυχούν οι εγώ θα ήθελα αυτές τις εικόνε που είδαμε σήμερα να τι μοιραστούμε με όλους τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου. Γιατί όταν ακούω ορισμένες από τις παρεμβάσεις, όταν άκουσα ορισμένε από τις παρεμβάσει στην ε, συζήτηση για το καλέ ε, στην Ολομέλεια εχθέ, ορισμένων συναδέλφων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μειοψηφία, καλό θα ήταν να τους ε, ταρακουνήσουμε λίγο αν θέλετε δείχνοντάς τους αυτές τις εικόνες. Θέλω να σας συγχαρώ για τη δράση σας, για το έργο σας. Και σας κυρία Δήμαρχε και ε, τους δύο εκπροσώπους της Ιταλικής Εκτοφυλακής και τον υπεύθυνο της επιχείρησης ε, Σοφία. Ε, αποτελείται παράδειγμα προς μνήμηση και για εμάς, ε, τους πολιτικούς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, γιατί συχνά εσείς αποτελείτε αντικείμενο επιθέσεων, αλλά οι μαρτυρίες που μας μεταφέρατε, ε, αυτά που μας δείξατε, αποδεικνύουν ότι ακριβώς επειδή έχουμε την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη, θα έχουμε τη δυνατότητα ή μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες τραγωδίες στο ανθρωπιστικό επίπεδο και επίσης μας θέτεται ενώπιον των πολιτικών μας ε, ευθυνών. Πριν από 15 μέρες με τον κύριο Φίσα, με τον κύριο ε, ε, Ποντσερίνη είχαμε συναντήσεις στην Τινησία με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Λιβύη, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Τινησία ακριβώς επειδή δεν μπορεί να βρίσκεται στη Λιβύη εξαιτία του πολέμου που συνεχίζει να μένεται, ε, των τεράστιων ε, δυσκολιών. Διαπιστώνουμε ότι στη Λιβύη δεν υφίσταται κράτος δικαίου, δεν υφίσταται καν κράτος θα έλεγε κανείς και αυτό δημιουργεί τεράστιες ε, δυσκολίες. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να αναφέρει κανείς για την Συρία. Σήμερα πάλι συζητήσαμε το θέμα της Συρίας στην Ολομέλεια. Και επιπλέον οι χώρες της Αφρικής, το αναφέρατε και εσείς, όλο και ε, περισσότερο αυξάνεται ο αριθμό των ε, προσφύγων και μεταναστών που έρχονται από χώρες της ε, Αφρικής. Και μην ξεχνάμε και την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική από ένα δισεκατομμύριο σήμερα σε 1,5 δισεκατομμύριο σε 10 χρόνια, επομένως, το, μέχρι το 2050. Συγγνώμη. Επομένω, οι καταστάσεις που συνεχίζουν να υφίστανται με τις συγκρούσεις θα πρέπει να μας απασχολήσουν ως επίγουσες. Την... Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κιέν. Να ευχαριστήσω την Τζούζη Λικολίνη, τη δήμαρχο της Λαμπεντούζα και τους δύο ποναβάρχους, τον ναυτικού και της εκτροφυλακής. Και ως εισηγήτρια μια έκθεση για τη Μεσόγειο όπου στην Επιτροπή μας στην Λίμπε καταφέραμε να συζητούσαμε το θέμα αυτό με μεγάλη πλειοψηφία τον Απρίλιο. Κατάφερα να, να κάνω αυτή τη δουλειά χάρη και σε εσά, γιατί κάναμε πολλέ ε, αποστολέ, με πολλέ συναντήσει με την Δήμαρχο, την ακτοφυλακή, τον ε, αντινάβαρχο, συναντήσαμε τον ναυτικό και αυτό μας βοήθησε. Να επενθυμίσω λοιπόν αυτά τα γεγονότα εδώ, λέγοντα ότι για αυτά τα θέματα μίλησε με μια φωνή το Κοινοβούλιο για ένα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Άκουσα την, την Δήμαρχο αυτά που είπε, τα συγκινητικά λόγια. Ήδη από το 2013 τα λέμε αυτά. με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, προσπαθώντας να ενισχύσουμε τις δράσεις έρευνας και διάσωσης. Εμείς είμαστε περήφανοι για την δουλειά που κάνετε εσείς εδώ. Γιατί μέσω της δουλειά σας καταφέραμε να δώσουμε προβολή σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτά τα γεγονότα και η προβολή αυτή περιλάμβανε και τη δικιά σας τη συμβολή, με τις δικές σας προτάσεις. Και Πρόεδρε, κάνω μια έκκληση. Εμεί θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να ξεπεράσουμε του εγωισμού των χωρών μελών. Είναι συμπαγή στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Πρέπει όμω να εργαστούμε ακριβώ για να ενισχύσουμε και την ευθύνη των υπολείπων χωρών μελών. Μόνο μια λέγια Ευρώπη μπορούμε να βγούμε από την κρίση και να δουλέψουμε πάνω ακριβώ στα βαθιά αίτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ε, παρουσία σας. Στον ΟΙΕ την περαισμένη εβδομάδα που είχα πάει, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ας πούμε ο Καναδάς δέχτηκε 35.000 ε, Σύριους και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούσαν καν να δεχτούν 5.000 από τις 160.000 καταστάση που είχαν υποσχεθεί πέρσι. Ούτε καν το μισό. Είναι δύσκολο λοιπόν να στήσουμε αξιόπιστα μια καινή προσπάθεια αν εμείς εδώ στην Ευρώπη δεν είμαστε σε θέση να δείξουμε και να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όπως έλεγε προηγουμένως η Σεσίλ, εδώ και καιρό ζητάει το Κοινοβούλιο ψηφίσματα τα οποία βασίζονται στην ίση κατανομή των ευθυνών μας που ήδη προβλέπουν οι συνθήκες μας, το 78 και 80 άρθρα της συνθήκης μας. Είναι, είναι γραμμένο αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό παραβιάζουμε τις συνθήκες μας. Και είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς και υπάρχει άλλο πρόσωπο της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει το πρόσωπο το δικό σας, αυτό που κάνουν τις ε, διασώσεις, που σώζουν ζωές. Και το καλύτερο πρόσωπο της Ευρώπης είναι οι οικοσαϊτείς, οι εθελοντές που προσπαθούν να συμβάλλουν με μια ελάχιστη ανθρωπιά και ανθρώπινη υποδοχή για αυτούς τους ε, μετανάστες και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η Ευρώπη με εσάς. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ένα τόσο περίπλοκο φαινόμενο δεν μπορούμε να το λύσουμε άμεσα. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, η οποία όμως βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να ενισχύει τη παρέμβαση στην θάλασσα και να οδηγήσει μεγαλύτερη ανταπόκριση από την Ευρώπη. Μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα και είμαι εισηγήτρια για τους ε, σοσιαλιστές για αυτό το θέμα, θα πρέπει να λύσουμε επιτέλους την υποκρισία της συμφωνίας του Δουβλίνου. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ασφαλείς διαδρόμους και να αποτρέψουμε τη διακίνηση ανθρωπίνων όντων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα βαθιά αίτια αυτού του φαινομένου με σωστές πολιτικές, εμπορικές, φορολογικές, εξωτικής πολιτικής ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή που ψεύσαμε χθε και τη ανισότητα, που είναι ένα κεντρικό ζήτημα της εποχής μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαράκα. Ευχαριστώ. Καλύτερα να το πω στα ισπανικά. Τα τελικά μου είναι της καταστροφής. Λέει ο κ. Μαραγκάλη. Εσείς είστε αυτοί που καλύτερα μας μεταφέρουν την πραγματικότητα που, τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζετε και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους πέρα από τα λόγια και πέρα από τη ρητορική. Τα δικά σας τα λόγια, κυρία Δήμαρχε, δεν ακούονται εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δύσκολο να ακούσει κανείς κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε τα γραφειοκρατικά, άλλη γλώσσα, αυτή δική μας. Εσείς μιλάτε Ιταλικά. Εσείς μιλάτε μια Ιταλική γλώσσα, γνήσια και βαθιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και ευχαριστώ για τα ειλικρινή σας λόγια. Να ευχαριστήσω και του εκπροσώπου ακτοφυλακή και του ναυτικού. Εσεί μα μεταφέρατε γνώση και συνέστημα και τα δύο. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Προκαλούν όμω απογοήτευση. Αν όχι εσεί, εμείς δεν θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε την απογοήτευση σε δράση, σε αποφασιστικότητα. Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε επανειλημμένο, νομίζω θετικά για αυτό το θέμα. Για το τι θα έπρεπε, τι θα μπορούσε να συμβαίνει στο θέμα αυτό. Πρόεδρε, ζητώ εσείς να αναλάβετε ένα γενικό ρόλο της Ευρώπης σε αυτό το ζήτημα και να καταλήξουμε σε μια πραγματική συναχία μεταξύ Κοινοβουλίου Δημάρχων, Κοινοβουλίου Πόλεων, Κοινοβουλίου Περιφερειών. Δεν είμαστε ως Κοινοβουλίο κατά της υποδοχής προσφύγων όπως λένε κάποιες χώρες μέλη. Απλά και μόνο δεν έχουμε εφαρμόσει ορατά και απτά τους μηχανισμούς που προβλέπονται. Τη στιγμή που η υποδοχή εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Και θα πρέπει ακόμα μετά από αυτά που ακούσαμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε Ονομοποιούμαστε ακόμα περισσότερο να το κάνουμε. Ας μην τους καλέσουμε να μην υποχρεώσουμε κανένα να δει το βίντεο που είδαμε στην αρχή. Αλλά σε όλα τα δημόσια σχολεία θα πρέπει να προβληθούν αυτά τα θέματα και στις αρχές, στις δημόσιες σε διάφορες χώρες. Και έτσι μόνο θα μπορούσαμε να αλλάξουμε επιτέλους την ευαισθησία που έχουμε για αυτό το θέμα. Η καλύτερη απάντηση στο δημοψήφισμα της Ουγγαρίας της Κυριακής είναι ακριβώς αυτή η συμμαχία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαίων πολιτών που ακριβώς περιλαμβάνει αυτά που είπατε και εσείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας και να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Νικολίνη και τους ε, ε, υποναπάρχους για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα, κλείνοντας τη συζήτησή μου, όχι μόνο να σας ευχαριστήσω, αλλά να σας μεταφέρω και κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, να πω ότι δεν θα είχα αντίρρηση ο κύριος Μελώνε την παρουσίαση του και ε, το βίντεο του να τα παρουσιάσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων. Äh. Νομίζω ότι έτσι να ευαισθητοποιηθούν θα είναι και ο κύριος Όρμπαν για παράδειγμα παρόν. Και θα πρέπει να δει τις διαστάσεις του προβλήματος και να καταλάβει περί τίνος μιλάμε. Τα αριθμητικά που, στοιχεία που μας δώσατε, αλλά και οι άνθρωποι που έχετε σώσει, πόσο μάλλον ε, οι νεκροί. Μόνο με έναν τρόπο που να τα περιγράψει κανείς αυτά, πρόκειται για ανθρωπιστική καταστροφή. Και μάλιστα, σε μια χρονική στιγμή που εσείς ε, κάνετε ένα ανθρωπιστικό μεγαλούργημα. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Ο καθένας που θα δει το βίντεο αυτό και όπως σας είπα είχα την ευκαιρία με την επιχείρηση Μαρενόστρουμ να δω επιτόπου ε, τους ανθρώπους σας. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς με λόγια. Ούτε στην ταινία φαίνεται αυτό. Θα πρέπει κανείς να το δει στην πραγματικότητα, να καταλάβει για τι δράμα μιλάμε. με την Τζούση και άλλους υψηλούς εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, βρέθηκα στην πρώτη επέτειο της καταστροφής της Λαμπετούζα. Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει κάτι τόσο τρομερό. Αλλά να μην σας κρύψω το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα κοινοβούλιο όπου υπάρχουν ευρωβουλευτές που μίλησαν για ανθρώπινα απορρίμματα όταν είδανε την εικόνα του μικρού αγοριού που, ε, είχε, τον οποίο είχα παρασύρει τα κύματα στην, στην ακτή του Μποντρούμ. Και δεν σας το λέω επειδή εδώ μας ανησυχεί αυτό, διότι εδώ πρόκειται για μειοψηφία, μία που φωνάζει όλο και πιο δυνατά, αλλά παρόλα αυτά μειοψηφία. Αλλά να μην αυταπατώμεθα όλο και περισσότερο υπάρχει αυτή η νοοτροπία και αυτή η ρητορική. Και να σας ε, πω ότι δύο Ιταλοί πολιτικοί που εδώ το γραφείο τους ε, έχουν που έχουν πει ότι όταν ε, βλέπω αυτά τα πράγματα θα ήθελα ε, να ακούσω κανόνια. Ε, πρόκειτο για τον επικεφαλής της Λίγα Νόρτ. Ο Φώση. Ο Ομπέρτο Μπόση, συγγνώμη. Εμείς ε, δεν ακούμε κανόνια, βλέπουμε το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό που ε, σώζει τους ανθρώπους αυτούς. Ε, είμαστε περήφανοι για σας εδώ στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό που ήρθατε εδώ σήμερα. Μία παρατήρηση για το Δουβλίνο. όταν διασώζεται τους ανθρώπους, όταν φτάνουν στο νησί της Τζούζα Νικολίνη, όταν ε, καταχωρίζονται στα Μητρώα, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Θα πρέπει η Ιταλία να εντάξει του ανθρώπου αυτού στην κοινωνία. Αλλά ξέρω, όλοι ξέρουμε ότι η Ιταλία δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη τη. Ούτε η Γερμανία δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη τη, Ούτε η Ελλάδα μπορεί να υποδεχθεί μόνη τη όλου αυτού του μετανάστε. Ούτε καν η Ιταλία, η Γερμανία και η Ελλάδα μαζί δεν θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών. Έτσι λοιπόν δεν χρειαζόμαστε το Δουβλίνο, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Και το α και το ω της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου θα είναι να έχουμε δίκαιο μηχανισμό κατανομής στην ε, Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε ενιαίες διαδικασίες αναγνώρισης, ε, πρότυπα για τους ανθρώπους αυτούς, διότι Αλλιώς θα γονατίσουν οι χώρες που πρέπει να φέρουν το βάρος αυτό. Αυτό ισχύει και για την Ιταλία. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας το 2015 ε, υποδέχτηκε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που είναι η μεγαλύτερη και η πιο πλούσια χώρα. Νομίζω ότι πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα της Γερμανίας. Είμαστε Γερμανοί. Ε, ε, είμαστε περήφανοι εμείς οι Γερμανοί για αυτό. Όμως, Εάν μοιράσουμε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες σε 508 εκατομμύρια, τότε δεν θα είναι πρόβλημα αυτό. Ο κάθε δήμαρχος που θα υποδεχτεί κάποιους ε, μετανάστες θα μπορέσει να τους ε, εντάξει. Εάν όμως ένα εκατομμύρια ε, πρέπει να ε, ε, πάνε σε μία χώρα ή δύο εκατομμύρια να πάνε σε τρεις χώρες, είναι αδύνατο αυτό. Είναι λοιπόν ευρωπαϊκό πρόβλημα το μεταναστευτικό, γι' αυτό χρειάζεται και ευρωπαϊκή λύση. Και πρέπει στο Κοινοβούλιο να καταβάλουμε ακούραστες προσπάθειες και δεν θα πρέπει να αποτύχει το ε, εγχείρημα αυτό λόγω του εγωισμού των κρατών μελών. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την ε, Τζούζα Νικολίνη, ε, και τους ε, κυρίους ε, που ήρθατε εδώ, αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά σας. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που αντέξατε το σύνορα. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά και τους διερμηνείς για την υπέρβαση του χρόνου. Ευχαριστώ.